Die Sitzung Συνεχίζεται η συνεδρίασή μα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι στη διάθεσή σα. Υπάρχουν αντιρρήσει, ενστάσεις. Δεν υπάρχουν. Κυρώνονται τα πρακτικά λοιπόν αυτά. Ναι. Μια αναγγελία, αγγελία Πρόεδρου.